και θα ήθελα σε όλες και όλους αλλά και ιδιαίτερα στις, στους γιώδεις τη της ομάδας να καταστήσω σαφές ότι τη Δευτέρα αυτή θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την έκθεση και τη συζήτηση με όλες τις πολιτικές πτυχές της όσον αφορά την ουσία όχι όσον αφορά τα άθρα που αναφέρονται στην επιτροπολογία γνωρίζετε ότι χθε ήταν 1η Δεκεμβρίου και επομένως αρχίζει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Άρα πάλι με τη σειρά τους όλα τα άρθρα της Επιτροπολογίας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Επ' αυτόν εργάζεται τώρα η νομική υπηρεσία αλλά και οι υπηρεσίε των χωρών μελών. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε λοιπόν εν προκειμένου. Άρα θα ε, συμφωνήσαμε ήδη με την Σουηδική Προεδρία ότι τα πολιτικά τμήματα όπου μπορούμε να συμφωνήσουμε αυτά να τα ολοκληρώσουμε και το τμήμα της Επιτροπολογίας να το διαπραγματευτούμε πλέον με την Ισπανική Προεδρία. Έτσι θα εξελιχθεί και το τεχνικό μέρος των διαπραγματεύσεων. Θα έχουμε δηλαδή τις ε, διαπραγματεύσεις για την Επιτροπολογία και μετά παρακαλώ οι σκιώδεις ηγητές να μεταβούν στις πολιτικές ομάδες και να συζητήσουν το θέμα και το αποτέλεσμα με τις πολιτικές ομάδες. Θα ήθελα να μιλήσω και με τον κύριο Κάπουλα Σάντος ή τουλάχιστον να με ακούει ο κύριος Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ. Είστε και εσείς ε, παρόν στις και γι' αυτό χρειάζομαι και τη συνεργασία σας. Παρακαλώ λοιπόν τους και οδησίγητες την Δευτέρα μετά από τον επίσημο τριμερή διάλογο να παραμείνουν λίγο στην αίθουσα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και μετά να πάνε στις πολιτικές τους ομάδες και μέχρι την Πέμπτη να δώσουν είτε σε μένα είτε στην γραμματεία της Επιτροπής το OK για τα θέματα τα οποία θα έχουμε ολοκληρώσει. έτσι ώστε και ο πρόεδρος της Επιτροπής να μπορέσει να συντάξει επιστολή προς τη Σουηδική Προεδρία για τα θέματα αυτά. Τότε μπορεί πλέον η Σουηδική Προεδρία αλλά και εμείς να βγει και να πει ότι μάλιστα αυτά τα ζητήματα ολοκληρώθηκαν, η συζήτησή τους ολοκληρώθηκε και βέβαια μένει πια το θέμα της επιτροπολογίας θα αρχίσει να συζητείται από τον Ιανουάριο με την Ισπανική Προεδρία. Γιατί μόνο όταν θα έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση των θεμάτων αυτών μπορούμε να το συζητήσουμε και να ψηφίσουμε πλέον στην Ολομέλεια. Αυτό θα είναι βέβαια μάλλον Ιανουάριο, όχι Ιανουάριο, Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Για όλους τους μετέχοντες είναι σημαντικό αυτό το πρώτο μέρος που έχουμε διαπραγματευτεί με τους Σουηδούς να το ολοκληρώσουμε. Δεν θέλουμε να αρχίσει και, νέα, και νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Προσπάθησα λοιπόν να σε εξηγήσω με ακρίβεια Είμαστε και εμείς κάπως σαν ένα πειραματόζωο τώρα γιατί είμαστε στη μεταβατική περίοδο ανάμεσα στην παλιά συνθήκη και στη νέα συνθήκη και είμαστε και η μόνη επιτροπή που έχει μια ψηφισμένη έκθεση και την οποία συζητεί με την Προεδρία του Συμβουλίου. Όλες οι άλλες εκθέσεις οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την ενδιάμεση ε, περίοδο βρίσκονται ακόμα ενώπιον των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Μόνο η δική μας έκθεση βρίσκεται εδώ. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι να προσέξουμε πολύ για, τα, για το νομοτεχνικό μέρος και όπως σας εξήγησα να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Γιάκλε για την παρουσίασή σας και να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Evans. Thank you. Um, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Γέγκλε για αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε, για τις ε, συναντήσεις, για τους σκιώδεις συγκητές και για το προσωπικό, για όλους δηλαδή που συμμετέχουν στις συζητήσεις. Και έχουν γίνει πολλές συνεδριάσεις και πολλές πληροφορίες ε, έχουν δοθεί τις τελευταίες ημέρες ε, προετοιμάζοντας τις συνεδρίες της επόμενης Δευτέρας. Πρέπει να σας πω όμως, εξ ονόματος των Πρασίνων, ε, ε, και της ομάδας μας δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής βεβαίως υπάρχουν πολλά θετικά σημεία μας, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το άρθρο 15 για παράδειγμα ε, για τη διαγραφή της παρέκκλησης καθώς επίσης και ορισμένα άλλα σημεία όπως ανέφερε και η ίδια η κυρία Γέγκλε αλλά αυτή η διαδικασία θα πρέπει να καταλήξει ε, σε ισχυρότερη νομοθεσία για την κατάσταση των ζώων, να υπάρξουν νέε μέθοδοι αντικατάσταση και διαρκώ βελτίωση όσον αφορά ε, τα πρότυπα της φροντίδα. Και ένα βασικό ζήτημα για μα είναι το άρθρο 2α έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για το ζήτημα αυτό ε, και ε, ακούστηκαν και απόψεις ε, νομικής φύσεως. Χαιρόμαστε όμως, λυπούμαστε όμως για τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να εγκρίνουν υψηλότερα πρότυπα. Δεν μιλώ μόνο για διατήρηση υψηλότερων προτύπων. Το επιχείρημα έχει να κάνει με την εναρμόνιση. Πάντως εμείς πιστεύουμε ότι όσο περνά ο καιρό, τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι σε θέση να θεσπίσουν καλύτερα πρότυπα, εάν το επιθυμούν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα για την ομάδα μας, διότι δεν ενθαρρύνει την εναρμόνιση προς τα πάνω, αλλά προς τα κάτω. Και στην ουσία ε, έχουν το πλεονέκτημα τα κράτη-μέλη με τα χαμηλότερα πρότυπα. Όσον αφορά το άρθρο 8 ε, για ε, ε, τα πειράματα στα, ε, στους πυθίκους. Ε, και εδώ ε, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και είμαστε απογοητευμένοι γιατί προτείνεται ο έλεγχος σε 25%. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Και όσον αφορά τη θεματική αναθεώρηση, εδώ θέλουμε μια πιο λεπτομερή παράγραφο όσον αφορά τη θεματική αναθεώρηση. Είναι πολύ κρίσιμη σημασία το ζήτημα αυτό για το μηχανισμό συμμόρφωση. Κάθε τέσσερα χρόνια δεν είναι και υπερβολή. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία εμπλέκονται ε, και τα θέματα δημοσίου ε, ε, και το γεγονός ότι το κοινό ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα ζητήματα αυτά θέλουμε πολύ συγκεκριμένους στόχους για την εισαγωγή νέων μηχανισμών αντικατάστασης για τα πειράματα. Έχουμε λοιπόν διάφορα προβλήματα με το κείμενο ως έχει, αλλά βεβαίως ε, θα ε, συμμετάσχουμε στη συνεδρίαση τη Δευτέρα ε, και συζητήσουμε με την κυρία Γέγκλε και θα κάνουμε τις παρατηρήσεις μας. Σίγουρα λοιπόν θα το συζητήσουμε με την ομάδα και θα σας δώσουμε την θέση μας την άλλη εβδομάδα όπως άλλωστε ζήτησε και η parole. Ευχαριστώ κύριο Καπούλα Σάντος, έχει δει το λόγο. Eh, σας ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γέλμπες, Γέγκλες, σας ζητήσω συγγνώμη, σας ζητώ συγγνώμη γιατί δεν πρόσεχα. Ένα, για ένα λεπτό αφαιρέθηκα, ξεκαθάρισα κάτι με τη γραμματεία. Ξέρω ότι εργαστήκατε πολύ σκληρά και η εργασία σας είναι εξαιρετική. Άλλωστε μας έχετε συνηθίσει εδώ και πολλά χρόνια σε τέτοια αποτελέσματα. Και σημειώθηκε πολύ μεγάλη πρόοδος χάρη στη δική σας συνεργασία. Από την άλλη μεριά, θα ήθελα να δικαιολογήσω την απουσία του σκιώδη εισηγητή γιατί στη Ρουμανία ε, βρίσκεται στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν θα είναι και την επόμενη εβδομάδα, θα είμαι παρόν για να, βρούμε, για να βρούμε μια λύση. Στην πολιτική μου ομάδα εξακολουθούμε να έχουμε κάποια προβλήματα, πάντως θα καταβάλουμε προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια λύση όσον αφορά το θέμα των ελέγχων, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, ελπίζω ε, να συμβάλλω ουσιαστικά για να εξακολουθήσουμε να σημειώνουμε πρόοδο. Και να σας πω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις προτάσεις και στην εργασία της κυρίας Γέγκλε και νομίζω ότι θα μας οδηγήσει σε αίσιο πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καπούλα Σάντος. Για ένα λεπτό δεν ακούστηκε η γαλλική μετάφραση, η διερμηνία προς τα γαλλικά, αλλά ελπίζω ε, να καταλάβατε όλοι τι έγινε στη συνέχεια. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Πάουλσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο περιλαμβάνει δύο πράγματα. Αφενός από αυτήν <clears throat> αποδείχθηκε ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του σχεδίου και δεύτερο σε σχέση με το σχέδιο της Κομισιόν Έχει αποδυναμωθεί σημαντικά η προστασία, της, ε, η των ζώων. Αφού η κίνηση, η μετακίνηση έγινε μάλλον υπέρ της έρευνας και της βιομηχανίας. Εν τέλει δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο κείμενο της Κομισιόν. Κάτι που θα ήθελαν οι πράσινοι και το καταλαβαίνω αλλά δεν είναι δυνατόν πλέον ούτε καν νομικά. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιστρέψουμε στην αρχική αυτή θέση της Κομισιόν. Μόνο συμβιβασμό μπορούμε να επιτύχουμε. Γιατί στην ψηφοφορία, στην Ολομέλεια, απορρίφθηκε ένα μέγα μέρος της εκθέσεως. Ελπίζω ότι αυτό θα μπορέσουμε να το αντιληφθούμε και να αντιληφθούμε επίσης ότι είναι σχετικά δυσχερής η θέση της κυρία Γέγλε. Έχουμε προσεγγίσει το Συμβούλιο πάντω. δηλαδή δεν μένουν τόσο κρίσιμα αποφασιστικά θέματα. Έχουμε φτάσει σε θέμα διατυπώσεων περισσότερο. Και γι' αυτό, όπως πίστευα και από την αρχή, μπορούμε όντως να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που να είναι λογικός για όλους. Δηλαδή σε μια νομοθετική ρύθμιση που να εξυπηρετεί και την έρευνα και τη βιομηχανία αλλά και τις που να είναι και αποδεκτή από τις ε, ομάδες προστασίας των ζώων που έχουν θεμητά ενδιαφέροντα και αυτές. εφόσον ε, κάποιοι θεωρούν ότι σε εγκαταστάσει έρευνα συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν ε, είναι σωστά, πρέπει να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνει και να διενεργεί ελέγχους. Αυτό θα έχει μεγάλη ωφέλεια για τις ε, οργανώσεις προστασία των ζώων, διότι τους ανοίγεται η νομική δυνατότητα να επικαλούνται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη ζητούν να διεξάγει ελέγχους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ντές έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την Ελίζα Πετιέγκλη για την εργασία που κατέβαλε σε αυτό το πολύ δυσχερές θέμα. Εγώ είμαι αρκετά χρόνια ευρωβουλευτής και το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι πάντα υπάρχουν τεράστιε αποκλήσει απόψεων για την προστασία των ζώων. Ποτέ δεν θα μπορέσει να βρει κανεί μια ρύθμιση που να ικανοποιεί όλε τι πλευρέ. Οι προστάτε των ζώων θέλουν πάρα πολύ αυστηρέ διατάξει. Οι ερευνητέ θέλουν περισσότερε ελευθερίε. Θα παρακαλέσω λοιπόν και εγώ με τη μου να καταλήξουμε κάποτε να εξευρεθεί ο συμβιβασμό, διότι α μην λησμονούμε ότι Ακόμα και αν εδώ στην Ευρώπη εφαρμόσουμε πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές, δεν σημαίνει ότι σε άλλα μέρη του κόσμου δεν θα γίνονται έρευνες με πειραματόζωα. Αν διώξουμε την έρευνα από την Ευρώπη, θα πάνε σε χώρες όπου δεν υπάρχουν κανόνο, καθόλου διατάξεις και δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των ζώων με τον τρόπο αυτό. Ας βρούμε λοιπόν ένα συμβασμό που να ικανοποιεί λίγο πολύ όλους. και να μπορούμε κι εμείς να εποφελούμαστε από έρευνα που να γίνεται με σωστό τρόπο. Ελπίζω όλες οι πολιτικές ομάδες να μπορέσουν να υποστηρίξουν εν τέλει την, ε, το αποτέλεσμα του συμβιβασμού που έχει διαπραγματευτεί η κυρία Γέγκλε. Ευχαριστώ κύριε Τέσ και τώρα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Κυρία Σουσάνα Λούμις Ευχαριστώ. Σύμφωνα με την έκθεση, του εισηγητή, είχαμε πολύ χρήσιμες διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι έχετε κάνει μερικές προσπάθειες για να επιτευχθεί λύση. Συζήτησαμε βεβαίω και με το Συμβούλιο και θα λέω ότι και εκεί επικρατεί το ίδιο πνεύμα. Φυσικά εκκρεμούν ορισμένα ζητήματα, αλλά από ό,τι βλέπω είναι κρίσιμα για την προστασία των ζώων και ελπίζω θα μπορέσουμε να τα ρυθμίσουμε για να επιτύχουμε ακριβώς συγκυρασμό όλων των συμφερόντων, όλων των πλευρών. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσει να συνεχίσει η Κομισιόν να διαδραματίζει ρόλο διαμεσολαβητή και να συνεισφέρει με τη γνώση που έχει ώστε να επιδεχθούν και οι απαραίτητοι συμβιβασμοί. Ευχαριστώ κύριε μου. Ο εισηγητή, μήπω θέλει να παρέμβει. Η κυρία Γέγλε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, ευχαριστώ τους και οδησηγητές καθώς και τους άλλους συναδέλφους. Αυτό που είπε ο Άλμπερτ στο τέλος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι τα πιο σημαντικά. Εάν καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, σε κάποια αποτελέσματα που θα καταστήσουν αδύνατο το έργο της έρευνας και της βιομηχανίας, θα σηκωθούν να φύγουν από την Ευρώπη. Και αυτό δεν εξυπηρετεί ούτε και τα ζώα, ούτε και τον κλάδο. Άρα, πρέπει να βρούμε κάποια ισορροπία για την πρόοδο και σε ό,τι αφορά την προστασία των ζώων και σε ό,τι αφορά του άλλους φορείς, έρευνα, βιομηχανία κλπ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας. Ασφαλώς υπάρχει δυνατότητα βελτίωση σε ορισμένα θέματα. Κύριε Κάπουλα το θα χαρώ πολύ να σας δω την Δευτέρα. Θα μπορέσουμε να ζητήσουμε τους ίδιου ελέγχου όπω αυτοί τους που επιβάλλονται στους ε, αγρότες. Και αυτό ήταν πάντοτε που ζητούσα εγώ. Πάντως, η έλεγχη είναι σημαντικό πράγμα και εφόσον οι έλεγχοι λειτουργούν, αποδίδουν και γίνονται και απροειδοποιητά, έχω την ελπίδα ότι θα ε, είναι επαρκής η προστασία των ζώων. Είναι σημαντικός στόχος αυτός. Άλλο σημαντικός στόχος για μας ως Επιτροπή και το βλέπουμε και στην έκθεση πρωτοβουλία τη κ. Πάουλσεν για την καλή μεταχείριση των ζώων. Σε τρία-τέσσερα χρόνια μπορούμε να ξαναρωτήσουμε μια έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Ποιε ήταν οι εξελίξει, αυτό μπορούμε να ρωτήσουμε τότε. Τώρα, οι χώρε μέλη, για παράδειγμα η Γερμανία, μπορούν να θεσπίσουν και υψηλότερα πρότυπα. Δεν προβλέπεται περιορισμός εξίσωση των προτύπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου καθίσταται απαραίτητο μπορούν να διατηρηθούν υψηλότερα στάνταρ. Επίσης, ξέρω ότι λαμβάνετε πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα, πολλά ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και εγώ το ίδιο. Μερικά είναι τέτοια που μπορούν να σας στερήσουν και τον ύπνο σας τη νύχτα. Εγώ καταφέρνω και κοιμούμαι ακόμα τη νύχτα. Πάντω εύκολη δεν ήταν η έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στον, στο επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων. Σχετικά με τη διαδικασία προπολογισμού 2010, την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο ξεκίνησε την συνδιαλλαγή με το Συμβούλιο. Η συγκεκριμένη είναι και πάλι η κυρία Γιάγκλη, η οποία θα μα παρουσιάσει το θέμα. Κυρία Γιάγκλη. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή σε σχέση με την προηγούμενη είναι απλώς αναψυχή, διότι <clears throat> το μόνο που ασχολεί εδώ είναι τα νούμερα και όχι τα συναισθήματα. Και επειδή ως Επιτροπή Γεωργίας επιτύχαμε πολλά στις διαπραγματεύσεις και ο προϋπολογισμός είναι <clears throat> πλέον έκθεση που εντάσσεται στη συναπόφαση. Στις 2 Σεπτεμβρίου διεξήχθη ψηφοφορία εδώ για τον αγροτικό προϋπολογισμό του 2010 στις 29 Σεπτεμβρίου διεξήχθη η ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και μπορέσαμε εκεί να περάσουμε όλες τις τροπολογίες μας, μεγάλη επιτυχία και στις 22 Οκτωβρίου έγινε η ψηφοφορία στην Ολομέλεια όπου με τη βοήθεια του Σούριαν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών πάλι μπορέσαμε να επιτύχουμε πολλά. Στις 18 Νοεμβρίου έγινε η συνδιαλλαγή μεταξύ Συμβουλίου ε, Κομισιών και Κοινοβουλίου. Ως εισηγήτρια για τον αγροτικό προϋπολογισμό ήμουν παρούσα στις συνδιαλλαγές και μπόρεσα να προβάλλω τις θέσεις μας. Τα πιο σημαντικά θέματα για μας είναι η έγκριση της ε, τροποποιητικής επιστολής υπαριθμών 2 της Κομισιόν για την κατηγορία 2 58,2 εκατομμύρια για α, πληρωμές, 64 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Σε σχέση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού για μέτρα παρεμβάσεως ανέρχεται κατά 415,4 εκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό ποσό είναι αυτό. Τώρα το Ταμείο Γάλακτος, όπως θέλετε πέστε το, ε, ε, δεν με ενδιαφέρει, αλλά έχουμε εκεί 300 εκατομμύρια ευρώ. Θα θυμάστε ότι τον Σεπτέμβριο η Επίτροπος εδώ είχε πει ότι δεν πρόκειται να δώσει ούτε μία δεκάρα. Μετά από τις πρώτες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο καταφέραμε να τις αποσπάσουμε 280 εκατομμύρια. Και τώρα εγώ επέμεινα τόσο πολύ, στήλωσα τόσο πολύ τα πόδια, όπου τελικά πέτυχα 300 εκατομμύρια. Καμιά φορά λοιπόν αποδίδει το να είναι κανείς ξεροκέφαλος. Θα μου πείτε τώρα τα 20 εκατομμύρια άξιζαν τον κόπο να γίνει ο καυγάς. Άξιζαν, διότι μπόρεσε να περάσει τις θέσεις της Επιτροπή Γεωργίας και το Κοινοβούλιο. Η ανάπτυξη τώρα της υπαίθρου 388 εκατομμύρια. Χρήματα για το γάλα στα σχολεία ανεβαίνουν κατά 7 εκατομμύρια και φτάνουν τα 76. Το προσχέδιο προϋπολογισμού ίσως πρέπει να το υπενθυμίσω, σε όλα αυτά τα κονδύλια επαναποκαθίσταται, ακόμα και σε αυτά που δεν ανέφερα πριν. Δηλαδή, περνούν όλα τα κονδύλια του αρχικού του προσχεδίου προπολογισμού συν τα ποσά που ανέφερα. Τα πιλωτικά προγράμματα δεν ήταν θεμελιώδε θέμα για την συνδιαλλαγή. Θα ψηφιστούν σε δεύτερη ανάγνωση. Άλλωστε δεν είναι υποχρεωτικέ δαπάνε και το Κοινοβούλιο έχει πια εκεί τον τελευταίο λόγο. Και γίνεται η ψηφοφορία, άλλωστε μάλιστα τώρα αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή προπολογισμών. Έχουμε 380 εκατομμύρια ε, περιθώριο για έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν τα επόμενα χρόνια, το χρόνο μάλλον. Αυτό μπορεί και να μεταφερθεί, μπορεί και να διατεθεί για υγειογικές δαπάνες εφόσον καταστεί απαραίτητο. Μπορεί όμως να πάει και σε προγράμματα συγκυρίας. Ο αγροτικός προϋπολογισμός του 2010 είναι 59,7 δις ευρώ στην κατηγορία 2. Και καταφέραμε ο δικός προϋπολογισμός φέτος να μην μειωθεί. Τα χρήματα που θα δοθούν στους αγρότες για την επόμενη χρονιά είναι εξασφαλισμένα. Στην ε, κατηγορία 2 δηλαδή, για θέματα που έχουν σχέση με αγορά και ανάπτυξη της υπαίθρου, αλληλεία, περιβάλλον, για το 2010, εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τον Δεκέμβριο στην δεύτερη ανάγνωση στο Στρασβούργο τα ποσά αυτά, εν τέλει τότε ο προπολογισμό μας θα έχει αυξηθεί κατά 9 δις σε σχέση με το 2009. Αυτό είναι και το κεντρικό εν τέλει μήνυμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω συνάδελφο να θέλει το λόγο. λόγος στην Κομισιόν λοιπόν, την οποία εκπροσωπεί η κυρία Μπόκμαν.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 E σας ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, με τον κίνδυνο να χαρακτηριστώ φαν της κυρίας Γέγλε, ε, συμφωνώ απόλυτα και, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά τα συμπεράσματα αυτά όσον αφορά ορισμένες από τις μάχες αυτές. Μάχες που κράτησαν μήνες, να μην σας πω χρόνια όπως για παράδειγμα το Ταμείο για το Γάλα. Ε, την, ε, την πρώτη μάχη την ξεκίνησε η κυρία Γιέγκλη για πριν πολύ καιρό. Για άλλη μια φορά λοιπόν τη συγχαίρω για την εξαιρετική της εργασία. Και ελπίζω και του χρόνου τα, τα αποτελέσματα είναι τέτοια μέσα με φέτο. Ο στην Κομισιόν. Πρόεδρε. Υπάρχει πλέον συμφωνία, όντως. Πρέπει να λάβει κανείς, μάλιστα υπόψη ότι χρειάστηκε να βρούμε χρηματοδόμηση από το δεύτερο πρόγραμμα ανάκαμψης. Καταφέραμε να πετύχουμε λοιπόν συμβαστική λύση. Είμαστε λοιπόν στα συν 420 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα ανάκαμψης, το οποίο ήταν ένα θετικό αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη της Κομισιόν, είναι ευτυχής εξέλιξη. Ότι για τα γαλακτοκομικά έχουμε 300 εκατομμύρια πλέον, το οποίο σημαίνει όμως ότι αφαιρέθηκαν 20 εκατομμύρια από τις εξαγωγικές επιτροφές για το γάλα. Και έτσι, στην τροποποιητική επιστολή, επελήθηκαν αυτές οι εξελίξεις. Να προσέξετε παρακαλώ ότι περιθώριο ήταν 500 εκατομμύρια, γιατί είχαμε περικοπές από την εκαθάριση λογαριασμών, όπως είχε προτείνει το Συμβούλιο, και αυτό συμπεριλήφθη στην συνδιαλλαγή έως το ποσό των 230 εκατομμύριων. Προβλέπονται δηλαδή αρνητικά έσοδα 230 εκατομμύριων πάνω από αυτά που είχε προβλέψει λοιπόν η Κομισιόν. Το έσοδο αυτό δεν είναι πραγματικό. Την τρύπα λοιπόν αυτού του προπολισμού πρέπει να γεμίσουμε. Τώρα το περιθώριό μας είναι 505 εκατομμύρια και η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί το κενό αυτό στον προπολισμό αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για έκτακτες ανάγκες όπως είπε και η κυρία Γιαγκλή, η συγγητρία. Εν τέλει λοιπόν ήταν θετικό το αποτέλεσμα για τη Γεωργία αλλά και γενικότερα ήταν καλό αποτέλεσμα το, για τη χρηματοδότηση του πρόγραμματος ανάκαμψης. για ε, σχόλια παρακαλώ ενδεχομένω. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Ευχαριστώ και όλες και όλους τους συναδέλφους και τον κ. Κάπουλα Σάντος βεβαίως είμαι ευγνώμων για κάθε φανατικό οπαδό. Αλλά εδώ με υποστηρίξαν και οι σοσιαλιστές και άλλες πολιτικές ομάδες γιατί το βασικό πρόβλημα εδώ για μας είναι να περάσουμε τα θέματά μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και να έχουμε και εκεί είχαμε μάλλον ευρεία ε, υποστήριξη από άλλες πολιτικές ομάδες και γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο σημείο, το οποίο είναι έκθεση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής, κοινωτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Η κυρία Μαρία Ντοσέου Πατράου Νέβες είναι η συντάκτρια της γνωμοδότησης. Στόχος της ε, ανακοίνωσης είναι προφανώς η πρόληψη των καταστροφών, μεγάλη σημασία στο θέμα, ιδιαίτερα για τον τομέα της γεωργίας. Η κυρία Πατράου Νέβες. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, προεδρεύοντα κυρίες και κύριοι ε, και τους υπόλοιπους προσκεκλημένους που ε, θα ήθελα να σας καλημερίσω όλους. Λοιπόν, το θέμα το οποίο μας απασχολεί σήμερα το οποίο θα το παρουσιάσω σε γενικές γραμμές, είναι η κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών καταστροφών ή ε, ανθρωπογενών καταστροφών. Δεν είναι ε, καινούριο θέμα. Είναι κάτι το οποίο απασχολεί ε, την, ε, μας απασχολεί εδώ και καιρό. Και είναι θέμα το οποίο αφορά άμεσα την Επιτροπή μας. Πρέπει να σας πω ότι η Επιτροπή μας ήδη συζήτησε το ζήτημα αυτό σε, με ευρύ τρόπο και συστηματικό. Και όλα αυτά κατέληξαν το Μάιο 2006 σε μία έκθεση. και βεβαίω ε, είχε γίνει και εργασία και σε άλλε επιτροπέ, όπω για παράδειγμα στην Επιτροπή περιφερειακή ανάπτυξη και στην Επιτροπή περιβάλλοντο. Το θέμα λοιπόν ε, προκύπτει εκ νέου και έρχεται στο προσκήνιο διότι ακριβώ πιστεύουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο εξακολουθεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε ε, λίγο ακόμα περισσότερα, να μην σας πω πολύ περισσότερα από ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, λάβουμε υπόψη μα αυτέ τι δύο παρατηρήσει, να σα πω το εξή. Ένα από του βασικού λόγου για του οποίου το θέμα μα απασχολεί εκ νέου είναι σίγουρα το γεγονό ότι οι φυσικέ καταστροφέ όχι μόνο αποτελούν μέρος της καθημερινής μας πρακτικής, αλλά όλο και ε, παρουσιάζονται μεγαλύτερη συχνότητα λόγω και της αλλαγής του κλίματος τα τελευταία χρόνια. Οι κλιματικές αυτές αλλαγές δείχνουν φάνηκαν ε, ακόμα περισσότερο μέσα από αυτά τα φαινόμενα ξηρασίας και υψηλότερων θερμοκρασιών σε χώρες του Νότου και βεβαίω αυτέ οι συνθήκε οδηγούν σε μεγαλύτερη εμφάνιση πυρκαγιών. Ταυτόχρονα είχαν πολύ περισσότερε βροχέ στι χώρε του Βορρά, με αποτέλεσμα πολύ περισσότερε πλημμύρε. Εδώ λοιπόν μιλάμε για την πρόληψη φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών. Δυστυχώ ε, το θέμα της κλιματικής αλλαγής θα εμφανίζεται διαρκώς στο προσκήνιο. Και πέραν των υποδείξεων, των προηγούμενων υποδείξεων, είδαμε και συστάσεων, είδαμε ότι ούτε καν αυτές δεν εγκρίθηκαν και δεν προτάθηκαν. Άρα πρέπει να αναδιατυπωθούν, γιατί πραγματικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ολέθρες συνέπειες αυτών των φαινομένων. φαινόμενα ε, τα οποία συνδέονται άμεσα με τις, ε, με τις αλλαγές του κλίματος. Γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα με την πρωτοβουλία του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, κοινοτική θέση ε, για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών και γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η αποφασιστική ε, στάση να υπάρξει τελικά και επιτέλους ένα ε, κοινοτικό μοντέλο αντιμετώπισης των καταστροφών και πρόληψή τους. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτό το χρόνιο πρόβλημα. Δηλαδή, απέναντι σε ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές στα κράτη-μέλη, πάντα προσκρούμε στο πρόβλημα ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές. Αν όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ένα σύστημα αυτόματης εφαρμογής απέναντι στις φυσικές καταστροφές, όχι μόνο η εργασία μας θα ήταν πιο αποτελεσματική, αλλά θα, θα ε, αφαιρούσε και μέρος ανησυχίας που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί, για παράδειγμα. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε με λεπτομέρειε ποια είναι η πρόθεση σε νομοθετικό επίπεδο τη Επιτροπή σε σχέση με την ανακοίνωση αυτή. Προσωπικά πιστεύω ότι η ανακοίνωση τη Επιτροπή για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών δεν ε, ε μας ε, δημιουργεί μια συγκεκριμένη εικόνα για το τι προθέσεις έχει σε νομοθετικό επίπεδο η Επιτροπή. Και αυτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε και ένα προσανατολισμό για να δούμε πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Και επίσης, να σας πω και το εξή. Βλέπουμε ότι η ανακοίνωση αυτή δεν περιέχει καινοτόμες προτάσεις σε σχέση με το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Δεύτερον, πολλές από τις προηγούμενες υποδείξεις και συστάσεις δεν εγκρίθηκαν όπως σας είπα. Σα παραπέμπω για παράδειγμα στην έκθεση του κυρίου Καπούλα Σάντο για, φυσικές καταστροφές, για, για τι φυσικέ καταστροφέ και τη γεωργία. Τρίτον, αυτή την ανακοίνωση την εξετάζουν διάφορε επιτροπέ μα. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε από ποια σκοπιά εμεί θα το δούμε το ζήτημα. Μετά από αυτέ τι γενικέ παρατηρήσει, θα ήθελα να σα πω το εξή. Βεβαίω, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα και θα ήθελα να σα πω το εξή. Μέσα σε ποια λειτουργικά όρια ε, θα ε, εφαρμοστεί, αν θέλετε, αυτή η ανακοίνωση. Γιατί, θα σας παραπέμπω στον τίτλο. Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Ποιε είναι οι φυσικέ καταστροφέ που θα πρέπει να μα απασχολήσουν. Μερικέ φορέ έχουν να κάνουν ε, με το κλίμα. Ξηρασία, για παράδειγμα, έχουμε εμεί ε, ε, πυρκαγιέ, χαλάζι, παγετό, πλημμύρε. Αλλά θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σεισμού, που, πλημμύρες που συνδέονται με τους σεισμούς κτλ. Καταλαβαίνετε δεν είναι όλα θέματα τα οποία αφορούν τη γεωργία. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να επιλέξουμε ορισμένες από τις φυσικές καταστροφές, εμείς από τη δικιά μας τη σκοπιά. Δηλαδή να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στις φυσικές καταστροφές που έχουν άμεσες βλαβερές συνέπειες για τη γεωργία. Μετά έχουμε τις ανθρωπογενείς καταστροφές. Και εδώ για να δούμε τι έχουμε. Πάλι πυρκαγιές αλλά με την έννοια του εμπρισμού ή σε ένα γενικότερο επίπεδο όλα τα φαινόμενα τα οποία μπορεί να οφείλονται στη μεταβολή του κλίματος που είναι ανθρωπογενής καταστροφή. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε, το δούμε ευρύτερα το ζήτημα ή πιο συγκεκριμένα να δούμε τα σημεία τα οποία αναφέρει και η ίδια ανακοίνωση Δηλαδή, εμείς πρέπει να δούμε, κατά την άποψή μου, την επίπτωση των καταστροφών αυτών στη γεωργία και να δούμε αυτές τις καταστροφές. Γιατί οι άλλες επιτροπές καταλαβαίνουν θα δουν τα πράγματα από τη δική τους σκοπιά. Οπότε μπορούμε να αναρωτηθούμε για το εξή. Ε, ε, ε, ε, τι γίνεται με τις διάφορες νόσους, για παράδειγμα. Ε, και τις ασθένειες. Ε, πρέπει να τα δούμε και αυτά. Άρα ε, να προσδιορίσουμε πιο συγκεκριμένα το, τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Πέραν όμως τούτου, να μην ξεχνάμε ότι τα θέματα δεν εξαντλούνται απόλυτα στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Γιατί, γιατί ο τίτλος χρησιμοποιεί τη λέξη πρόληψη. Ενώ το κείμενο δεν, ανα, δεν αναφέρεται μόνο στην πρόληψη, αλλά και στην παρέμβαση, στην περίπτωση που ε, έχουμε τέτοιε φυσικέ καταστροφέ. Βλέπετε λοιπόν τι δυσκολία υπάρχει. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την πρόληψη από την αντιμετώπιση. Ο τίτλος λοιπόν είναι παραπλανητικός, κατά κάποιο τρόπο. Γιατί διαβάζοντα το κείμενο της Επιτροπής, βλέπουμε ότι δεν περιοριζόμαστε μόνο στην πρόληψη, αλλά φύγουμε και το θέμα της αντιμετώπισης και της ε, παρέμβασης. Οπότε θα έλεγα ότι ίσως θα πρέπει να αφήσουμε τις θεωρητικές παρατηρήσεις που ήδη έχουν γίνει και να μιλήσουμε για ένα πιο συγκεκριμένο μοντέλο και ένα σύστημα που θα δίνει απαντήσεις στις διάφορες καταστροφές που εμφανίζονται. Ένα πρότυπο το οποίο, ε, και ένα μοντέλο, ένα σύστημα το οποίο θα μπορούσε να εφαρμόζεται αυτόματα μόλις προκύψει μια φυσική καταστροφή. Και ανεξάρτητα με το σύστημα ή το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει ε, και, αν θα και, να ζητήσουμε επαρκή χρηματοδότηση για να μπορέσει να λειτουργήσει το σύστημα. Άρα υπάρχει και το θέμα της χρηματοδότηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα... Αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσε φορές το ακούμε τελικά τι θα γίνει. Θα αφορά πολύ συγκεκριμένου σκοπού, γιατί τότε αποκλείονται άλλε καταστροφέ με ολέθριες συνέπειες για τη γεωργία, όπως για παράδειγμα η ξηρασία. Επίσης δεν είναι ενδιαφέρον για μας, εάν δεν ε, περιοριστούμε μόνο στην πρόληψη και περάσουμε και στην παρέμβαση, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους γεωργούς. Ε, για παράδειγμα, ασφάλιση από ασφαλιστικές εταιρείες, ένα σύστημα ασφάλισης κοινό και για τα 27 κρατημέλη που να ασφαλίζει τους γεωργούς έναντι φυσικών καταστροφών. Κοιτάξτε, τόσα χρόνια έχουμε την ΚΑΠ και όμως δεν έχουμε σύστημα ε, κοινή παρέμβασης. Αν τα αφήσουμε όλα αυτά στα, χέρια των κρατών μελών και για την πρόληψη και για την παρέμβαση στο πλαίσιο των φυσικών καταστροφών και ε, ανθρωπογενών καταστροφών τότε θα έχουμε Μία Ευρώπη, έχει δύο, αλλά πολύ με ταχυτήτων. Μπορούμε να μιλήσουμε, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πολλή ώρα για το θέμα αυτό που μας απασχολεί. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση για τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν εδώ θα με βοηθήσει και εμένα για να δω προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθώ μετά από αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και έτσι ώστε να υπάρξει και μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων και στη συνέχεια να πάμε σε πιο συγκεκριμένου προσανατολισμού που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην αερογραμματότηση αυτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκαρθία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχει δίκιο η συγκήτρια. Κυρία Πατράου. Στο ότι η Επιτροπή μας πρέπει να απαντήσει από τη σκοπιά της υπαίθρου, της ε, γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Εγώ είμαι σκισκιώδη συγκήτρια στην Επιτροπή τη Ουσία, στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Και εκεί ε, τα πράγματα τελείω διαφορετικά. Και η σκοπιά είναι και τελείω διαφορετική, η προσέγγιση είναι διαφορετική. Εμεί λοιπόν πρέπει να συμπληρώσουμε ε, την έκθεση τη ε, Επιτροπή των Συναδέλφων και ε, Περιβάλλοντο. Και έχει δίκιο κυρία Πατράου. Το πιο, το πιο σημαντικό ζήτημα είναι ακριβώς να βρούμε λύσεις και πρόληψη. Νομίζω ότι ένα από τα πιο θετικά μέτρα σε επίπεδο πρόληψη των φυσικών κινδύνων για τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι ακριβώ να εστιάσουμε την προσοχή μας στον πληθυσμό ε, και στους, ε, στους, στους οικισμούς αν θέλετε. και, ως, και, και αριθμητικά οι γεωργοί αλλά και ως πυρήνες οικισμών, οικιστικοί πυρήνες θα πρέπει να μείνουν στην Ήπεθρο. Γιατί διαφορετικά εξαφανίζονται αυτοί που ε, διαφυλάσσουν την ύπεθρο, που είναι οι γεωργοί κτηνοτρόφοι. Ο Βοσκός που βοσκάει τα πρόβατά του ε, και που προειδοποιούσε στη Μεσογειακή Ευρώπη για το ότι υπάρχει μία πυρκαγιά τελικά αντικαταστάθηκε από νέου ε, που κάθονται και παρατηρούν ε, τα δάση και βλέπουν αν υπάρξει φωτιά. Μα καταλαβαίνετε ότι ε, με αυτόν τον τρόπο χάσαμε του τους βοσκούς και αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο τα απολέστηκαν θέσει εργασία, αλλά χάσαμε και του φύλακε του δάσου. Βεβαίω, έχει δίκιο. Η πρόληψη είναι το βασικό ζήτημα. Και αν λάβουμε υπόψη ποιε είναι οι, βασικέ φυσικέ βασικές φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη, θα έλεγα ότι έχουμε τρία είδη. Πυρκαγιέ, πλημμύρε και ξηρασία. Τρία αυτά είδη αυτή πρέπει να είναι και οι τρει ε, στόχοι ε, τη έκθεση κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι μια βασική πολιτική, ευρωπαϊκή, πραγματική, ολοκληρωμένη και για όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε ε, τη συζήτηση και να την αφήνουμε στα, κράτη στα, επιμέρους κράτη-μέλη. Δεν έχει νόημα 27 διαφορετικές πολιτικές υπέρ των δασών στην Ευρώπη Επίση, κοινοτική νομοθεσία για την καταπολέμηση των πυρκαγιών και τη ξηρασία. Για να βελτιστοποιήσουμε τα, μέτρα, τα μέσα τα οποία υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να γίνει με συντονισμένο τρόπο. Δεν μπορεί εμεί να κάνουμε κάτι και στην Πορτογαλία κάτι άλλο. Ε, εδώ μιλάμε για την Ιβερική Χερσόνησο, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι διαφορετικό στην Αυστρία ή στην Ιταλία. Εδώ μιλάμε για τι Άλπε. Και βεβαίω εδώ ε, ε, ε, συμπεριλαμβάνουμε και τη Γαλλία. Άλλο πρέπει να κάνουμε στην Ουγγαρία και άλλο στην Αυστρία. Μα όχι, όλοι μαζί πρέπει να κινηθούμε. Επίση πρέπει να υπάρχουν οι απαρκεί πόροι για να δοθεί μια ταχεία απάντηση σε περίπτωση καταστροφών. Σα μιλάω για την πολιτική προστασία. Και αυτό ε, θα πρέπει ε, ένα ε, ακόμα μέσον που θα πρέπει να συμπληρώσει τα μέσα τα οποία υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίω πραγματική και αληθινή υποστήριξη σε επίπεδο ενίσχυση. Και εδώ μιλώ για το Ταμείο Αλληλεγγύη. Μια μεγάλη, θαυμα, μεγαλειώδης ιδέα, θαυμάσια ιδέα. Αλλά κάθε καλοκαίρι. Περνάει το καλοκαίρι και κάθε Σεπτέμβρη γιατί μιλάμε. Ή για πλημμύρε ή για πυρκαγιέ. Ε, ας σταματήσουμε πια τις βλακίες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε έμβαση εκεί που πρέπει και αν είναι θέμα χρημάτων να ξεπεράσουμε αυτή την... Ε, ε, ε, αυτή τη στάση. Ε, ας σταματήσουμε να είμαστε ε, τσιγκούνιδες. Αν χρειάζονται χρήματα, ας τα δούμε και στα δώσουμε. Και θα πρέπει έτσι ε, να, να δώσουμε το μέσο αυτό σε αυτούς που πραγματικά το χρειάζονται. Επιτέλους. Αυτά ήθελα να πω και βεβαίω είμαι στη διάθεση τη κυρία Πατράου για να συνεργαστούμε και ελπίζω να έχουμε μια πραγματική έκθεση που να συμπληρώνει αυτήν τη ε, Επιτροπή Περιβάλλοντο, να έχουμε μια, ε, ε, μια έκθεση η οποία και σε πολιτικό επίπεδο και σε τεχνικό επίπεδο να είναι ε, προωθημένη στο βαθμό που πρέπει για να δοθεί απάντηση στα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ και την συγγετρία με αφορμή αυτά τα οποία είπε η κυρία Καρσία, χρειαζόμαστε πολιτική απάντηση Και υπάρχουν και άλλα θέματα. Στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή πληττόμεθα από σοβαρέ πλημμύρε σε διάφορα σημεία της χώρας. Και αυτοί που ξέρουν την περιοχή και την ιστορία ξέρουν ότι αυτό είναι χωρίς προηγούμενο, είναι απρόβλεπτο. Μπορεί να συνδέεται με την αλλαγή του κλίματος, όμως επιπλέον μπορεί να πηγάζει από έλλειψη πολεοδομίας, άγνοια των βασικών κανόνων στην κατασκευή αποστρακιστικών έργων, η επέκταση φυσικά των πόλεων επηρεάζει την ύπεθρο. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε προσεκτικά. Μίλησε επίσης με ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις αγρικίες τους λόγω Τη πλημμύρα και μα είπαν ότι δεν συντηρούνται κανάλια, αποστραγγιστικά έργα και ούτω καθεξή. Ακριβώς επειδή η υπέρμαχοι του περιβάλλοντο και οι γεωργοί βρίσκονται σε σοβαρή αντιπαράθεση και αυτή την αντιπαράθεση πρέπει να γεφυρώσουμε. Σε πολλέ δυστυχώς περιπτώσει αλλά και σε αυτήν την περίπτωση, ενώ με δίστανται σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ δηλαδή υπερμάχων του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινοτήτων και των αγροτών. Παλιά, ε, για παράδειγμα, γινόταν η συντηρήση των ποταμών και των καναλιών. Τώρα όμω, μόλις πάει κάποιο να αυξήσει την ε, ροή του νερού για να γίνει σωστά η αποστράγγιση, ε, αρχίζουν οι περιβαλλοντικές ομάδες να αντιδρούν. Άλλε φορέ δικαιολογημένα, άλλε όχι. Να το σημειώσουμε και αυτό, διότι τελικώς άνθρωποι χάνουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Αυτό συμβαίνει στην Ιρλανδία και σε άλλες χώρες όλο και περισσότερο. Οπότε περιμένω να δω ε, το, σχέδιο για να σχολιάσω περαιτέρω. Ευχαριστώ κύριε Καπουλεσάντος. Κύριε Καπουλεσάντος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είναι πάρα πολύ θετική αυτή η παρουσίαση στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε το θέμα αυτό χωρίς ε, να ε, μας πιέζουν τα γεγονότα. Θυμάμαι το 2006 ήμουν εισηγητής μετά από μια μαύρη χρονιά όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές που είχαν ε, γίνει. Πυρκαγιές, ε, τρομερές και από την άλλη ε, τρομερές πλημμύρες που είχαν ε, δημιουργήσει θύματα και είχαν προξενήσει μεγάλες καταστροφές στα κράτη-μέλη. Όταν λοιπόν κανείς είναι αγκασμένος να εργαστεί υποπίεση και να μιλά για μέτρα ε, που πρέπει να ακολουθηθούν, ε, τότε καταλαβαίνετε δεν είμαστε νυφάλοι, Η συζήτηση δεν γίνεται με νυφάλιο τρόπο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το ε, θέμα τη κοινοτική αντιμετώπιση, παρόλο πρέπει να πω ότι από το 2005 μέχρι σήμερα βεβαίω και υπήρξε πρόοδος. Δεν εδόθη συνέχεια σε ορισμένε προτάσει που κάναμε, αλλά σε άλλε εδόθη. Και να σα υπενθυμίσω, κυρίε και κύριοι, ότι στην, ε, ε, στον τελευταίο έλεγχο τη υγεία τη Γεωργία εξασφαλίσαμε να υπάρξει ένα κοινοτικό πλαίσιο ε, για το θέμα ε, των, ασφαλίσεων, για παράδειγμα. Δηλαδή, ήδη τα έχουμε συζητήσει αυτά. Και μερικέ φορέ, βεβαίω, όμω όλα αυτά ε, στην πράξη εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θέλω να υποστηρίξω την τοποθέτηση της εισηγήτριας, γιατί νομίζω ότι η έκθεση θα πρέπει να μιλά για την πρόληψη, αλλά κυρίως και πάνω απ' όλα να προτείνουμε μηχανισμούς παρέμβασης είναι πάρα πολύ σωστό να εντοπίσουμε τις αιτίες, να δούμε ποιες είναι φυσικές αιτίες και ποιες καταστροφές είναι ανθρωπογενής φύσεως. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν και εκείνες τις καταστροφές που έχουν άμεσα συνέβηση για τη Γεωργία, γιατί αυτό είναι η δική μας αρμοδιότητα και επίσης να πω και το εξή. Και απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτός ο κατάλογος των μέσων που είχε δεσμευτεί να μας παρουσιάσει το 2009 θα ήταν κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί θα μπορούσαμε να μάθουμε ακριβώς και να ξέρουμε ακριβώς τι νομοθετικά και χρηματοδοτικά μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Όλα αυτά θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα. Αυτός ο κατάλογος θα μπορούσε να χρησιμεύσει για να γνωρίζουμε τι μπορούν να μας δώσουν τα μέσα αυτά και τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, όσον αφορά ε, την υλοποίηση ενός συστήματος ασφαλίσεων, γεωργικών ασφαλίσεων. Σας παρέπεμψα στο θέμα του ελέγχου της υγείας, γεωργίας. Πάντως θα πρέπει να ξέρουμε πολύ συγκεκριμένα μέσα από αυτόν τον κατάλογο των μέσων και των εργαλείων ποια είναι αυτά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κάτω από ποιε συνθήκε. Αλλά επαναλαμβάνω, η πολιτική μα ομάδα και εγώ ίδιο είμαστε στη διάθεσή σα έτσι ώστε η έκθεση αυτή και αυτή η γνωμοδότηση να είναι χρήσιμη και να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Γεωργία και του Ευρωπαίου Γεωργού. Ευχαριστώ. Έχουμε και άλλους ομιλητές εδώ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι το έργο είναι πολύ σημαντικό εδώ, τόσο για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και δι των ανθρωπογενών. Ε, πρέπει όμως να μην ξεχνούμε και τις δύο πτυχές. Όσον αφορά τις φυσικές καταστροφές, μπορεί το θέμα του κλίματος και της ενδεχομένης αλλαγής του κλίματος να είναι σημαντικό, γιατί όντως δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται για μακροσκοπική, μακροπρόθεσμη αλλαγή του κλίματος. Πάντως έχουμε να κάνουμε εδώ με καινούργια φαινόμενα. Ε, έργα λοιπόν ότι έχουμε σίγουρα επιπτώσεις στην γεωργία. Και αυτό αφορά όλες τις χώρες που πλήττονται από την εξερασία. Σήμερα γίνεται σημαντική δουλειά από τους γεωργούς για να προσαρμόσουν τις ποικιλίε που σπέρνουν, για να τις προσαρμόσουν συγκεκριμένα σε ένα πιο ξηρό κλίμα. Πρέπει λοιπόν, σε επίπεδο έρευνας και με δημόσιους πόρους και σε συνεργασία με τους αγρότες να δομολογήσουμε συμμετοχική έρευνα για να επιταχύνουμε ακριβώς την προσαρμογή αυτών των νέων σπόρων στις νέες συνθήκες. Συνθήκες οι οποίες αφορούν την ξηρασία. Χρειάζεται λοιπόν έρευνα, χρειάζεται ενημέρωση. Πρέπει να προσαρμόσουμε τη γεωργία, όχι με το συνηθισμένο τρόπο, αλλά να υποφεληθούμε από τη δουλειά που κάνουν οι αγρότε για να τροποποιήσουν ακριβώ του σπόρου, να αλλάξουν του σπόρου το, ο καθένα στον τομέα του. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, όσον αφορά τι ανθρωπογενεί καταστροφέ. Μιλούμε μεταξύ άλλων για τι πυρκαγιέ. Εδώ και χρόνια πολλά. Ξέρουμε και λέμε ότι ένα καναντέρ είναι πολύ πιο ακριβό από έναν γεωργό είναι ένα βοσκό. Λοιπόν, Εμεί θέλουμε γερού και βοσκούς παντού. Χρειάζεται μια θετική πολιτική κινήτρων για να εγκατασταθούν στις ζώνες που κινδυνεύουν από την ξηρασία, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, γιατί ακριβώ μέσω του καθαρισμού που επιτυγχάνει μέσω τη κτηνοτροφία σε αυτές τις περιοχές μπορούμε να ελέγξουμε τις πυρκαγιέ. Δείτε τι γίνεται στα μεσογειακά δάση. Χρειάζεται διαχείριση. Διαχείριση όχι μόνο του χώρου εν αλλά ειδικά των δασών. Διότι τα δάση ανήκουν εν και στα ζώα. Χρειάζεται λοιπόν μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του δάσου. Το δάσο δεν υπάρχει όπου υπάρχει για να δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα. Είναι και ένα χώρο αναψυχή. για τι ανθρωπογενεί λοιπόν καταστροφές εφιστάμεθα όλοι τι επιπτώσει τη βιομηχανική γεωργία στην Βρετανία. Στην Βρετάνη, με συγχωρείτε. Στη Βρετάνη, ε, μεταξύ άλλων. Παρατηρούμε τον πληθωρισμό που συνιστούν τα ε, φύκια λόγω ακριβώ τη αυξημένη παρουσία νητρικών στην θάλασσα, λόγω υπερτροφισμού. Το φαινόμενο αυτό απαγορεύει την ύπαρξη οποιοδήποτε άλλου είδους ζωής. Καταστρέφουμε λοιπόν τα εδάφη, τις θάλασσες, εξαιτία ακριβώς των εκτατικών καλλιεργιών. Ο Στεφαν Λεφόλ ασχολείται με το θέμα. Το θέμα είναι να προλάβουμε ακριβώς τους κινδύνους στους οποίους συνεπάγονται οι εκτατικές αγροτικές πρακτικές. Ύστερα μιλάμε για πλημμύρες, αλλά να μην ξεχνούμε και την ε, το θέμα της αποστράγγισης. Το νερό πρέπει να κυκλοφορεί πιο γρήγορα για να αρδεύονται αυτές οι καλλιέργειες. Αλλά αυτό είναι μια τεχνητή κατάσταση. Έχουμε μεγαλύτερες κατασκευές, μεγαλύτερες υποδομές που αλλοιώνουν το τοπίο της υπαίθρου. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να σχολιάσουμε. Να πούμε δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές στην εκμετάλλευση της υπαίθρου. Αυτό είναι ένα τμήμα της πρόληψης ακριβώς των ανθρωπογενών κινδύνων. Ευχαριστώ. Κύριε Μπουβέ, δίνω τον λόγο στον κύριο Συρκεύσκη. Χρειαζόμαστε απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, οι οποίε θα επιτρέψουν στην Ένωση να δράσει ταχύτερα στην αντιμετώπιση των καταστροφών. Το Κοινοβούλιο και οι βουλευτές αυτό ζητούν. Οι πολίτε μας περιμένουν από εμά να κάνουμε κάτι και να αλλάξουμε τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτών. Πρέπει να δράσουμε λοιπόν τώρα και να περιμένουμε μήνες όπως συμβαίνει συνήθως. Δεύτερον, όσον αφορά τους τύπους των καταστροφών φυσικά έχουμε πλημμύρες αφενός Πιστεύουμε προκειμένου ότι περισσότερε επενδύσει θα μπορούσαν να προλάβουν αυτέ τι καταστροφέ. Οι επενδύσει αυτέ πολλέ φορέ καθυστερούν. Αδικαιολόγητα μάλιστα. Θα αντιμετωπίσουμε επίσης στο μέλλον πρόβλημα με το νερό. Χρειάζεται λοιπόν από σήμερα να επενδύσουμε μεγαλύτερους πόρους για να διαχειριστούμε το νερό καλύτερα. Πρέπει όμως να διαχειριστούμε και τους κινδύνους. Το συζητήσαμε αυτό ήδη, όμως οι ασφαλίσει δεν είναι λύση, γιατί συνήθω οι ασφαλίσει ε, ωφελούν μάλλον τι ασφαλιστικέ εταιρείε. Πρέπει τέλος να εξορθολογήσουμε τις περιβαλλοντικές μας παρεμβάσεις. Πολλές φορές περιβαλλοντικές ομάδες παγώνουν επενδύσεις, οι οποίες όμως είναι απολύτως απαραίτητες για να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες καταστροφές για παράδειγμα, η δημιουργία λεκανών σε ορισμένες περιοχές ή τη συγκέντρωση του νερού. Αποστραγγιστικά έργα. Κάποιες λύσεις από αυτές πρέπει να ενταχθούν τέλος στις μελλοντικές δημοσιονομικές πρόπτικες για να γίνουν και τμήμα της γεωργικής μας πολιτικής. Ευχαριστώ. Κύριε Πόλσον. Ε, Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ε, εγώ θα μιλήσω μόνο για τα δάση. Και θα τονίσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές είναι εξίσου σημαντικές με την ξηρασία σε όλη την Μεσόγειο. Και έχω στο μυαλό μου κυρίως ε, τον Νότο. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση η οποία απαιτεί αναπροσαρμογή των τρόπων δράσης. Τα πράγματα εξελίσσονται, οι τάσεις διαφαίνονται. Δεν έχουμε λόγο να περιμένουμε άλλο. Τα δάση στην πατρίδα μου, την Σουηδία, στην Φιλανδία, κινδυνεύουν, αλλά οι κίνδυνοι είναι διαφορετικοί από αυτούς που απειλούν τη Μεσόγειο. Βιολογικά, καταρχήν, τα δάση επιτελούν διαφορετική λειτουργία στον Βορρά και στον Νότο. Εμείς, για παράδειγμα, στον Βορρά δεν έχουμε καθόλου πυρκαγιές ή τουλάχιστον σχεδόν καθόλου πυρκαγιές. Αυτά. Ολόκληρη λοιπόν η συζήτηση για την πρόληψη των πυρκαγιών στα δάση στην περιοχή της Μεσογείου ε, βεβαίως είναι σωστή αλλά μας ε, ε, βγάζει κάπως από το σωστό δρόμο. Αν λάβουμε υπόψη ότι στο βορρά τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Βεβαίως υπάρχει η αρχή της αλληλεγγύης και όλοι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως θα πρέπει να ισχύει και να υπερισχύει η αρχή της ελεγγύης και βεβαίως ε, το κόστος πρέπει να το μοιραστούμε όλοι. η κατάσταση στις χώρες ε, ε, της ε, Μεσογείου δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί έχουμε τις καταστροφικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και όλοι θα πρέπει να λάβουμε την ευθύνη μας για το ζήτημα αυτό. Τώρα, δεν θέλω να πω με τι, τι ακριβώς πρέπει να περιέχει η γνωμοδότηση επιλέξει. να σα πω ότι στην Βόρεια Ευρώπη ε, το φαινόμενο ε, της πλημμύρας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και... Αν κάτσουμε να δούμε τι γίνεται και στο, στο βορρά της Ευρώπης θα δούμε ότι ε, πραγματικά ε, είναι, ε, ε δημιουργεί τρομερή εντύπωση. Ε, κατασκευάζονται σπίτια δίπλα στη θάλασσα. Γίνονται, ε, και όμως ξέρουμε όλοι τι ακριβώς γίνεται. Άρα πρέπει να κάτσουμε λίγο και να σκεφτούμε αφού υπάρχει κίνδυνο της πλημμύρας στη χώρα μου. Υπάρχουν οικισμοί, κοινότητες οι οποίες ασκούν τη χωροταξία, κάνουν, ρυθμίζουν τη χωροταξία και τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουμε κάποια θέση σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα πέντε ομιλητέ στον κατάλογο μου. Κ. Σέλβοτ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την έκθεση. Ευχαριστώ για τα σχόλια των συναδέλφων με τα οποία συμφερώ. Και με τόνισα ότι μεγάλες περιοχές της Ιρλανδίας, τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση είναι κάτω από το νερό αυτή τη στιγμή, πλημμυρισμένες. Και αυτό επηρεάζει το περιβάλλον, τις υποδομές, την ζωή των τοπικών κοινωνιών. Έχουν καταστραφεί ολόκληρε σοδιέ και παραλαμβάνω οι επιπτώσει στη ζωή των τυπικών κοινωνιών είναι τεράστιε. Ευχαριστώ πολύ για την συνδρομή του Ταμείου Λιλεγγύης. Πρέπει όμω για να είναι επαρκή η συνδρομή του τα κριτήρια να τροποποιηθούν και είναι σκόπιμο να συζητήσουμε το θέμα. Έχουμε μάλιστα μια έξοχη ευκαιρία εδώ να συζητήσουμε το αν η εκνηστέρων παρέμβαση είναι επαρκή. αντί για την πρόληψη μέσω αποστραγγιστικών έργων, για παράδειγμα, ε, μέσω της ε, αφαίρεσης ε, φρακτών και άλλων εμποδίων που χρειάζονταν στο παρελθόν, αλλά όχι σήμερα. Το θέμα είναι ότι η ελέγχη του κλίματος είναι πραγματικότητα. Είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε με τα συμπεράσματα. Στα τέλη Νοεμβρίου στην Ιρλανδία και αυτό ισχύει και την ε, Βρετανία, η βροχόπτωση αυξήθηκε κατά 10%. Αυτό θα συμβεί μάλλον και τον Δεκέμβριο και μιλάμε για μια αύξηση 20%. Πηγαίνουμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα στην ε, Κοπενχάγη για να μιλήσουμε για την αλλαγή του κλίματος. Πιστεύω ότι όλες οι επιτροπές, όχι μόνο η Επιτροπή Γεωργίας, να ενημερωθούν και να καταστρώσουν ένα συντονισμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Καλή λοιπόν η αντίδραση, αλλά πολύ καλύτερη η πρόληψη. Ευχαριστώ λοιπόν για την έκθεση. Περιμένω το τελικό κείμενο. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική έκθεση για το μέλλον και την ευημερία των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λάβαμε μέσα υπόψη και τις αλλαγές του κλίματος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλγουκ. Ο κύριος Χάουσλινγκ. Πρόεδρε, συμφωνώ με τα περισσότερα αυτά που ακούστηκαν. Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα. Νομίζω ότι δεν είναι και δυνατόν πάντοτε να διακρίνει κανείς ποιες είναι οι φυσικές και ποιες είναι οι ανθρωπογενείς καταστροφές, γιατί συχνά αυτά είναι τόσο στενά συνδεδεμένα. Για παράδειγμα, οι πλημμύρες. Πάντοτε μετά τις πλημμύρες αποδεικνύεται, για παράδειγμα, όπως είπε και κάποιος πριν, ότι οφείλεται στην υπερβολική αστική συγκέντρωση ή στις, στα πολλά κτίσματα ή ότι δεν πρέπει να ασφαλτοστρώνουμε ή να κλείνουμε με τσιμέντο ε, όπως στη Γερμανία κάθε μέρα, ε, κάθε μέρα 120 εκτάρια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό πρέπει να αρχίσουμε και ως Επιτροπή Γεωργίας να ασχολούμαστε κάποια στιγμή και με την προστασία του αγαθού γη, έδαφος. Όσο τα καταστρέφουμε περισσότερο, τόσο περισσότερες πλημμύρες και τα σχετικά προβλήματα θα αντιμετωπίζουμε. Άρα κάποια συμπεράσματα πρέπει να βγάλουμε εδώ και όχι απλώς προθέσεις και δηλώσεις προθέσεων. Τώρα για τις πυρκαγιές δασών. Το καλοκαίρι Πάντοτε και όλο και περισσότερες πυρκαγιές δασών διαπιστώνονται παντού. Όταν περάσει η μεγάλη εντύπωση από τα μέσα επικοινωνίας κλπ. όλοι τα λησμονούν και ξανά το επόμενο καλοκαίρι. Αναδάσωση είναι το θέμα εδώ. Γίνεται σωστή αναδάσωση, για παράδειγμα, ιδιαίτερα στις μεσογειακές χώρες και είναι επαρκής η επιτήρηση των δασών υπάρχουν συμπεράσματα που εξάγονται, πρέπει να εφαρμοστούν με συνέπεια. Και συνέπεια χρειάζεται και σε πολλά πράγματα, όπου επιτέλους κάποιος, ε, κανείς πρέπει να διαρωτηθεί πώς είναι δυνατόν να μην μπορούμε να ξεφύγουμε από τους φαύλους αυτούς κύκλους εφαρμόζοντας κάποια πράγματα. Ευχαριστώ. Κυρία Μάτια παρακαλώ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συμβάλλω σε αυτήν την συζήτηση σχετικά με τα δάση που άπτεται βεβαίω του περιβάλλοντος αλλά και τη γεωργίας. Να ευχαριστήσω καταρχήν την εισηγήτρια η οποία έλαβε υπόψη τη τα σχόλια περί δασοπονία. οπότε δεν περιτεύει να επανέλθω στο θέμα των δασών και της ξηρασίας, στα μέρα τα οποία σχολίασαν οι συναδελφοί μου. Όμως, τα θέματα των καταιγίδων πρόσφατα Γερμανία, Αυστρία, το εντενέθμα στην Γαλλία, είχαμε νεκρούς, στα νοτιοδυτικά επίσης πέρσι. Οι σειρές αυτές καταιγίδες οδήγησαν σε συζητήσεις περί της διαχείρισης των δασών. Εδώ μιλούμε βεβαίω για πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την διαχείριση των δασών κατόπιν αυτών των ε, ακραίων καιρικών φαινομένων. Ίσως λοιπόν μαζί με τους γεωργούς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για διαχείριση δασών. Γιατί αυτά που συνέβησαν στη Γαλλία συνέβησαν και στη Γερμανία. Θεωρώ λοιπόν ότι απαιτείται μια ευρύτερη συζήτηση προς θέματος. Οπότε, ρωτώ, με φορμή την έκθεση, να μιλήσουμε, μάλλον προτείνω για πρόληψη και βεβαίω για την ανταπόκρισή μας, τις επεμβάσεις μας με διάφορα εργαλεία μεταξύ των οποίων και το Ταμείο Αλληλεγγύης στην περίπτωση που συμβαίνουν αυτές οι καταστροφές. Ε, το τελευταίο ήταν κάτι το οποίο είχε μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο. Το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι βεβαίω ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινοτική προσέγγιση, αν θέλετε, είναι πολύτιμη για τους πολίτες μας, οι οποίοι πλήττονται από φυσικέ καταστροφές. Εγώ θυμούμαι στη Λορένη την φοβερή κοινή καταιγίδα ήταν τρομακτική η απογοήτευση με τα ξεριζωμένα δέντρα, τι διακοπέ ηλεκτρικού ρεύματο. Εκεί δεν επένευε κανεί, ούτε καν το Ταμείο Αλληλεγγύη. Ήμασταν μόνοι μα. Και βεβαίω μετά από λίγου μήνε αποκαταστάθηκε η κατάσταση, αλλά τότε μα είπαν η κοινότητα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αμέσω, τουλάχιστον για τι επόμενε εβδομάδε. Περιμέναμε μήνε. Αισθανθήκαμε μόνοι μα, απολύτω μόνοι μα, κύριε Πρόεδρε. Χρειάζεται λοιπόν να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και εκ των υστέρων έστω, να υπάρχει κοινοτική προσέγγιση, ε, αλλιώς νομίζω ότι κάνουμε λιγότερα από αυτά που είναι το καθήκον μας να κάνουμε. Ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Άγνιου. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν αυτές τις φοβερές λέξεις, κλιματική αλλαγή. Πολλές, αλλαγές, πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ λαμβάνονται με βάση τις κλιματικές αλλαγές. Τα στατιστικά στοιχεία των επιστημόνων για το φαινόμενο αυτό επίσης αναφέρονται. Εγώ ζω, μένω κοντά ε, στο Πανεπιστήμιο του East Anglia που είναι εξειδικευμένο σε θέματα μετεωρολογίας. Ίσως να γνωρίζετε αλλά και να μην γνωρίζετε ότι πριν από δύο εβδομάδες ε, διέρευσε το γεγονός ότι οι επιστήμονες αποκρύπτουν το γεγονός ότι στην ουσία μειώνονται οι θερμοκρασίες. Καταλαβαίνετε αυτό μπορεί να είναι και ποινικό αδίκημα. Οριζ... Την επόμενη εβδομάδα, μείνε από εσά θα πάτε στην Κοπεχάγη για να μιλήσετε για τι κλιματικέ αλλαγέ. Για καθίστε μια ή δύο μέρε για να, ε, για να πάτε ε, και σε μία άλλη συνδιάσκεψη με τίτλο Climate Sense, κλιματική λογική, για να ακούσετε και την άλλη άποψη. Ε, οι επιστήμονε που θα έρθουν σε αυτή τη δεύτερη συνδιάσκεψη είναι τόσοι πολλοί που θα κρατήσει δύο μέρε. Εσεί τώρα θα έχετε αρμοδιότητες συναπόφαση. Θα πρέπει λοιπόν να βασίζετε τι αποφάσει σα ε, όχι σε προπαγάνδα αλλά και σε ευσεβεί πόθους, αλλά σε πραγματικά επιστημονικά στοιχεία. Ευχαριστώ και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Αλμπερτέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στην κυρία Πατράων Νέβες για την εκπόνηση της έκθεσης. Πάντως για το θέμα αλλαγής του κλίματος πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γι' αυτό έχω ανοίξει και το κομπιούτερ μου εδώ. Βλέπω τα επίπεδα των πλημμυρών μιας μικρής πόλης στο Μάιν το Würzburg το 2003 μετρήθηκαν 153 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο. Βγήκαν οι εφημερίδες και είπαν τρομερή καταστροφή, φταίει η αλλαγή του κλίματος, φταίνε τα τσιμέντα που κλείνουν το έδαφος κτλ. την 21 Ιουλίου 1382, όπου πέρασαν τα διπλάσια κυβικά μέτρα, τριπλάσια κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Μα δεν υπήρχαν τότε ούτε ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε τίποτα. Και εκτός από τους κατοίκους του Βίλσπουρ, κανένας άλλος δεν έμαθε για την πλημμύρα. Και ακριβώς 100 χρόνια μετά, 1483, 250 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο και άλλα τέτοια 1562, 350 κυβικά μετά. Μα ποια ήταν, ποια ήταν τότε τα αίτια. Έφταιγε πάλι η σύγχρονη γεωργία, η αλλαγή του κλίματος. Μα πέρναγε το διπλάσιο και τριπλάσιο νερό τότε. Και θα μπορούσα να σας πω τα ίδια πράγματα και για το Δούναβι. Τα ίδια επίπεδα πλημμυρών από τον Μεσαίωνα και στο Δούναβι, όπως το Βέλσπρουκ. Ας είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί. Πάντοτε υπήρξαν αλλαγές του κλίματος. Μπορώ να σας βρω και στατιστικές ότι είχαμε και υψηλότερε διακυμάνσει θερμοκρασιών. Δεν προσπαθώ να εμφανίσω το πρόβλημα ως δίθεν κινδυνο, αλλά πολύ συχνά ορισμένοι κάνουν πολιτική business για τα πράγματα αυτά. Και σίγουρα θα χαρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες άμα ανέβουν τα ασφάλιστρα για πλημμύρε και καταστροφέ των σπιτιών. Τώρα, για τι πυρκαγιέ. Πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορούν να σβήνονται ταχύτερα οι πυρκαγιέ. Η πυρκαγιά του δάσου οδηγεί σε καταστροφή εάν δεν μπορέσει να σβηστεί έγκαιρα. Άκουσα ότι στην Ελλάδα, όπου είναι φοβερές οι πυρκαγιές, σε, ένα, σε μια χώρα με 11 εκατομμύρια ε, Κατοίκου έχουν 12.000 επαγγελματίες πυροσβέστες. Εμείς στη Βαβαρία, ε, στη, Βαβαρία έχουμε εθελοντές πυροσβέστες. Κάθε ένας που γίνεται 16 χρονών πηγαίνει στην ε, πυροσβεστική και γίνεται, μαθαίνει πυροσβέστης. Εμείς έχουμε 200.000 πληθυσμό και έχουμε πάλι 12.000 πυροσβέστες. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ξέρουν τι να κάνουν για να σβήσουν μια πυρκαγιά και σε ένα δάσος. Πρέπει να τα σκεφτούμε λιγάκι αυτά τα πράγματα. Μήπω και σε μια χώρα όπω η Ελλάδα ή άλλε, η Ισπανία ή η Πορτογαλία, να εισαχθεί ο θεσμό τη ε, εθελοντική πυροσβεστική, ίσω και με υποστήριξη τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για την τεχνική υποστήριξη, να υπάρχουν και τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Ε, μία από τι αιτίε όπου η πυρκαγιά του δάσους γίνεται καταστροφή είναι όταν δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι και αρκετά τεχνικά μέσα για να την αντιμετωπίσουν. Νομίζω καλύτερα να περιοριστούμε σε κάποια λογικά πράγματα και όχι να καθόμαστε να θρυνούμε γοερά για πράγματα τα οποία δεν ε, κάνουμε τίποτα για να σταματήσουμε. Και η Ευρώπη υποστηρίζει βέβαια τις χώρες μέλη για την βελτίωση της προστασίας κατά των πλημμυρών. Πάλι από την δική μου την περιφέρεια υπήρχε ένα μέρος όπου κάθε χρόνο γινόταν πλημμύρες και με σημαντική ενίσχυση από τις Βρυξέλλες έγιναν έργα τα οποία μάλιστα έχουν και οικολογικό χαρακτήρα και οι άνθρωποι δεν χρειάζεται πλέον να φοβούνται ότι θα πλημμυρίσουν τα σπίτια τους. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες, πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε ώστε να προχωρήσουμε λίγο σε αυτές τις υποθέσεις. Ας τα συζητήσουμε λοιπόν αυτά και με λίγο αντικειμενικό πνεύμα και όχι μόνο όπως μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κύριε Ντές και εγώ πιστεύω ότι αυτό το σύστημα των εθελοντών πυροσβεστών είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα μπορούσε να, θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή έμπνευση και για άλλα κράτη-μέλη. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λεφόλ. Ε, κοιτάξτε, να, θέλησα να πάρω το λόγο γιατί ξεκίνησε καλά θα έλεγα. Μιλήσαμε για την καταπολέμηση, για τον αγώνα κατά των φυσικών καταστροφών και βεβαίως ε, πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι φυσική καταστροφή και τι είναι ανθρωπογενής. Να απαντήσω στον κύριο Ντέσ και στον κύριο Άγνιου. Η Βαβαρία είχε καλυφθεί από 100 150 μέτρα στην εποχή των παγετώνων. Η Σαχάρα ήταν ε, τροπική ζώνη. Κοιτάξτε, ε, πάντα υπήρχαν οι κλιματικές αλλαγές σε πλανητική κλίμακα. Αυτό μας εμποδίζει να σκεφτούμε τις συνέπειες που συνδέονται άμεσα κύριε Ντες στο γεγονός ότι ε, απορρίψαμε στην ατμόσφαιρα αυτό που για 100 εκατομμύρια χρόνια αποθήκευε ε, στη γη η φύση. Τώρα, οι κίνδυνοι συνδέονται με τις αλλαγές, βεβαίως. Εμείς ως πολιτικοί πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε τους κινδύνους και κατά πόσο μπορούμε να τους περιορίσουμε. Μα αυτό είναι το θέμα της έκθεσης, αν δεν κάνω λάθος. Για του εθελοντέ πυροσβέστε έχουμε πολλού στη Γαλλία. Είναι πολύ καλό το σύστημα, αλλά αυτό νομίζω ότι ισχύει και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Τώρα, να βοηθήσει η Ευρώπη για να προχωρήσουμε περισσότερο, βεβαίω. Η διαχείριση των δασών με διαφορετικό τρόπο σήμερα ε, πρέπει να γίνεται με πιο παγκόσμιο τρόπο ή τουλάχιστον σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Συμφωνώ. Ε, γιατί αποθηκεύει τον άνθρακα ε, και αποτελεί ένα δομικό ε, στοιχείο του, του, του χώρου το δάσος. Βεβαίως και το ξέρουν και οι χώρες του Βορρά. όταν κανείς ε, στη Φινλανδία και δει ότι οι λίμνες αναλλάσσονται με τα δάση, καταλαβαίνει περί τίνο πρόκειται βεβαίω. Επανερχόμαστε στη ζήτηση σαν να κάνουμε τώρα ε, μία αντιπαράθεση για την ε, ε, υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό είναι ένα θέμα. Βεβαίω έχουμε την θέρμανση του πλανήτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένε απαντήσει. Και σωστό, αναφέρεται και στα αρχή τη έκθεση. Τι να κάνουμε για να περιορίσουμε του κινδύνου που προέρχονται από τι φυσικέ καταστροφέ. Αυτή είναι η αρμοδιότητά μα, αυτή είναι η ευθύνη μα και εδώ πρέπει να σταθούμε. Ευχαριστώ. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Εκάουτ. Πρόεδρε. Κάθε φορά που τα θέματα άπτονται της αλλαγής του κλίματος, όλοι συζητούν πολύ προθυμία, αν όντως υπάρχει ή όχι. Λοιπόν, όσον αφορά το σχολείο του κυρίου Άγνιου και το αν πράγματι συμβαίνει αλλαγή ή όχι, ε, εκατοντάδες επιστήμονες Ισχύζεται ότι όντω συμβαίνει. Λοιπόν, εγώ δουλεύω για το θέμα εδώ και χρόνια, γνωρίζω του ανθρώπου στο Πανεπιστήμιο East Anglia ε, που ασχολούνται με την αλλαγή του κλίματο και αν θέλετε, φέρτε του εδώ να σα πούν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Λέει ο κ. Σάγνιο ότι ε, χαίρεται που στην Κοπενχάγη θα ευχαριστούν άνθρωποι που υποστηρίζουν δεν συμβαίνει η αλλαγή του κλίματος. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι για την Κοπεχάγη. Είναι ευχή ότι υπάρχει. Ε, θα προσταθεί και μία μέρα στο πρόγραμμα. Θα πρέπει εβδομάδε ενδεχομένω να προσταθούν. Αλλά στη φάση αυτή, για την έκθεση τουλάχιστον, δεν έχει και μεγάλη σημασία να συζητήσουμε εδώ εάν συμβαίνει η αλλαγή του κλίματο ή όχι. Υπάρχουν, και θα υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι δεν συμβαίνει. Πάντω, σίγουρα, ακόμη πιο σίγουρα, κάποιοι υφίστανται ήδη τι επιπτώσει τόσο από φυσικέ όσο και από ανθρωπογενεί καταστροφέ. Και αυτό είναι το αντικείμενό μα εδώ. Πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτέ τι καταστροφέ. Λοιπόν, να συζητήσουμε στη συνέχεια και για την πρόληψη και μετά για την αντιμετώπιση. Από την πλευρά τώρα των Γεωργών, γιατί είμαστε Επιτροπή Γεωργία εδώ, και όχι Επιτροπή Περιβάλλοντο, θέλουμε να εξετάσουμε τον ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει η Γεωργία στην πρόληψη και στην προσαρμογή. Ένα από τα βασικά θέματα εδώ είναι η πολύ λειτουργική, αν θέλετε, γεωργία. Γιατί αν δούμε με τον παραδοσιακό τρόπο την γεωργία, πολύ δύσκολα θα αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές της μεν και της δε. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα προσέγγιση να εμβαθύνουμε δηλαδή σε όλες τις διαφορετικές λειτουργίες της γεωργίας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι καταστροφές και αφήνοντας τους επιστήμονες ε, να συζητήσουν το κατά πόσο πρόκειται για φυσικέ Η κυρία Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα παρακαλέσω να πάρουμε πολύ στα σοβαρά τη συζήτηση αυτή και με κανένα τρόπο να μην θεωρήσουμε το θέμα ανώδυνο βλέπω ότι διαγράφεται ένα σημαντικό κίνδυνο εάν αρχίσουμε τώρα να μην παίρνουμε στο σοβαρά τις υποθέσεις αυτές. Έχουμε στο μεταξύ βάσεις επιστημονικών δεδομένων στις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε και στην ομόσπονδη χώρα μου, Σλέσβι Χόλσταϊν, ζούμε ανάμεσα σε δύο μεγάλες θάλασσες και βλέπουμε να πληθαίνουν οι θύελες αλλά και να ανεβαίνει και το επίπεδο της θάλασσας. Και εάν κάνουμε τις προβολές, αν δεχτούμε τις προβολές που κάνουν οι επιστήμονες, θα μειωθεί, θεωρούμε ότι θα μειωθεί η ε, χώρα μας κατά το 1 τρίτο του έδαφος της τα επόμενα 50 χρόνια. Άρα λοιπόν ας επανέλθουμε σε μια αντικειμενική συζήτηση και ας αφήσουμε τα σκιάχτρα να δούμε όλοι που βρίσκονται οι ευθύνες μας να εξετάσουμε τα επιστημονικά δεδομένα και να δούμε ποιου νέου δρόμου μπορούμε να ακολουθήσουμε. Η αύξηση του διοξιδίου του άνθρακου στα τελευταία χρόνια οφείλεται στι δικέ μα δραστηριότητε. Δεν θυμούμε η γιαγιά μου να είχε αυτοκίνητο, ούτε θυμούμε η γιαγιά μου να χρησιμοποιούσε σπρέι για τα μαλλιά. Α είμαστε λοιπόν λίγο πιο αντικειμενικοί, Α σταματήσουμε να παριστάνουμε ότι δήθεν αυτά είναι σενάρια τρόμου που ε, είναι για να φοβήσουν τον κόσμο και να ψάχνουμε να βρούσουμε στατιστικές πριν από αιώνε. Βεβαίω και τότε υπήρχαν φυσικέ καταστροφέ. Αυτά που βλέπουμε όμω σήμερα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην τεχνική εξέλιξη που έχει σημαντικέ επιπτώσει στη φύση. Ευχαριστώ πολύ κύριε μου και με συγχωρείτε και πάλι για το λάθος μου προηγουμένω. και που σαν το τελευταίο ομιλητή. Ε, ένα μεγάλο ποσοστό των ε, πυροσβεστών μας και στη χώρα μου την Πορτογαλία, πάνω από 90% είναι εθελοντές. Υπάρχουν και επαγγελματίες πυροσβέστες. Αυτοί είναι κατεστημένοι σε ορισμένες μεγάλες πόλεις της Πορτογαλίας. Εγώ έγινα μάρτυρας των μεγάλων ε, πυρκαγιών του 2005 για όσους δεν ζουν στο νότο της Ευρώπης είναι δύσκολο να φανταστούν μέσα σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου και να ξεσπούν τέτοιες πυρκαγιές. Και να μην υπάρχει ούτε σταγόνα βροχής στον ορίζοντα και ακόμα και οι ακτίνες του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές με βαρύτατε ε, συνέπειες. Τέτοιε τραγωδίες και μετά από τις τραγωδίες αυτές καλούμαστε να ε, βελτιστοποιήσουμε πολλούς μηχανισμούς. Λαμβάνονται μέτρα, ε, αγοράζονται αεροσκάφη πυρόσβεσης, αλλά όσα μέσα και να υπάρχουν, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές έγκαιρα και με τρόπο αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση. Ίσως να μην εκφράστηκα καλά περιορίστηκα ε, για το θέμα της πυροσβεστικής στην Ελλάδα γιατί με σώπαρε πραγματικά μια χώρα που έχει περίπου 12 εκατομμύρια κατοίκους να έχει μόνο 12.000 πυροσβέστες. Βρίσκω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ λίγοι. Τέτοιες καταστροφές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τόσο ε, περιορισμένο προσωπικό. Αυτό το στοιχείο μου το έδωσε μια Ελληνίδα συνάδελφός μου, ότι έχουν μόνο 12.000 ε, πυροσβέστες. Έχουν βέβαια πολλά πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά δεν έχουν επαρκές προσωπικό εδάφος. Εγώ πάντως θεωρώ ότι πρέπει να λαμβάνουμε όλα τα μέτρα πρόληψης, όλα τα δυνατά μέτρα πρόληψης, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι. Το μόνο που είπα είναι ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι ποτέ δεν υπήρξαν αλλαγές κλίματος στην ιστορία. Και εγώ προσπαθώ να δώσω το καλό παράδειγμα. Εδώ και χρόνια έχω κάνει ε, πολύ καλές ε, μονώσεις στο σπίτι μου. Έχω αλλάξει την παλιά μου ε, θέρμανση, τον παλιό μου καυστήρα που έχει και πετρέλαιο και χρησιμοποιώ τώρα έναν που χρησιμοποιεί ρινίσματα ξύλου. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε και αυτές τις πτυχές και να μην παριστάνουμε. Ε, πράγματα. Θα κερδίσουμε την υποστήριξη των ε, ανθρώπων τότε περισσότερο εάν προσφέρουμε λύσεις και όχι εάν τους τρομοκρατούμε. Ευχαριστώ. Λόγω στην Κομισιόν. Η πείτε από τον κύριο Κρίστοφερ Άλλην σήμερα. Πρόεδρε, Καταρχήν ένα ευχαριστώ από την Κομισιόν για το ότι το Κοινοβούλιο ανέλαβε την πρωτοβουλία να συντάξει αυτή την έκθεση για το σημαντικό θέμα της πρόληψης των καταστροφών. Εμπλέκονται προκειμένου διάφορες επιτροπές, το οποίο αντικατοπτρίζει τη σημασία την οποία αποδίδει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας στο θέμα. Λίγα λόγια για το παρελθόν. Να εξηγήσω πώς φτάσαμε στην ανακοίνωση. Το 2008 η Κομισιόν ενέκρινε την ανακοίνωση περί της αντιμετώπισης των καταστροφών, στην οποία λέγαμε ότι χρειάζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος, της διαχείρισης δηλαδή των καταστροφών με έμφαση στην πρόληψη και βεβαίως την αντιμετώπιση και την αναδιάρθρωση. Εστιάσαμε στη συνέχεια στην πρόληψη, γι' αυτό και η Κομισιόν το 2009, τον Φεβρουάριο συγκεκριμένα, ενέκρινε την ανακοίνωση για την κοινοτική προσέγγιση περί προλήψεως φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Συνεπώς, περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον και τη δική σας συνεισφορά περί πρόληψης. Η θέση μας είναι ότι υπάρχουν εργαλεία και μηχανισμοί με τη μορφή οδηγιών, για παράδειγμα, που ασχολούνται με την πρόληψη. Υπάρχει οδηγία για τις πλημμύρες, για παράδειγμα. Υπάρχουν όμως και χρηματοδοτικά εργαλεία μέτρα πρόληψη μπορούν να χρηματοδοτηθούν βάσει της περιφερειακής πολιτικής, στο πλαίσιο τη γεωρικής πολιτική και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει και η ίδια η Κομισιόν πιστεύει ότι η, απόσπαση, ή, προσέγγιση είναι αποσπασματική και ότι πρέπει να ιδρύσουμε μια ενιαία προσέγγιση για να τα ενσωματώσουμε όλα αυτά σε μια ενιαία προσέγγιση για να έχουμε αποτελεσματική πρόληψη. Γιατί αποδίδουμε τόση σημασία στο θέμα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι του. Στη δεκαετία του 90 συνέβησαν περίπου 100 καταστροφές λόγω δυσμενών κυρικών συνθήκων. Στη δεκαετία του 2000 έφτασαν ήδη τις 150. Αυτή είναι η πρόκληση που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Στην ανακοίνωση, στην έκθεση μάλλον προτείνονται διάφορα βήματα. Τομείς στους οποίους πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο. Γνωρίζουμε την κατάσταση. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι περισσότερο στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε καταρχήν να ενισχύσουμε αυτά τα οποία, να βελτιώσουμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε για το πρόβλημα. Αναπτύσσουμε επίσης μεθόδους ανάλυσης κινδύνου και κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπιση των κινδύνων σε περιφερειακό επίπεδο. Η Κομισιόν σκοπεύει να εκδώσει κατευθυντήριε γραμμέ που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να εντείνουν τι προσπαθίε του. Όσον αφορά την χρηματοδότηση, επειδή ακούστηκαν σχετικά σχόλια σήμερα, η Κομισιόν συμφωνεί ότι εν ώψη των δημοσιονομικών προοπτικών και τη έγκριση διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, καλό θα είναι να εστιάσουμε στην πρόληψη. Η Κομισιόν θα ακούσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι απόψει του Κοινοβουλίου στη φάση αυτή σχετικά με το τι μέτρα μπορούν να ληφθούν με τη χρηματοδότηση των κοινωτικών ταμείων, ώστε να χρησιμοποιήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κοινωτικά κονδύλια για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. Τέλος, ίσως θα ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με τις προθέσεις της Κομισιόν και το πού ακριβώ βρισκόμαστε. Η ανακοίνωση του 2009 προβλέπει συγκεκριμένα βήματα για μια νέα προσέγγιση των μέτρων πρόληψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σαφώ καταθέτουμε ένα σχετικό έγγραφο προς τα κοινωτικά όργανα να συλλέξουμε απόψεις και με βάση αυτό και με βάση τις υλοποίησεις των μέτρων που ήδη λαμβάνουμε, η Κομισιόν ενδέχεται να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες εφόσον παραστεί ανάγκη. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτά είναι συνακόλουθο της Λευκής Βιβλίου για την αλλαγή του κλίματος σαφώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των δασών, το οποίο έθιξαν διάφοροι βουλευτέ εδώ, και το με τη μορφή μια πράσινης βίβλου για την προστασία των δασών, που προβλέπεται να εγκριθεί από την Κομισιόν στις αρχές του 2010. Αυτό θα αποτελέσει και μια ευκαιρία να εξετάσουμε δελεχώ το θέμα των δασών και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένων βεβαίω των καταστροφών. Όσον αφορά τα μέτρα ανάκαμψη και αποκατάσταση, πολύ σημαντικά μέτρα εννοείται. Ε, εδώ εμείς περιλαμβάνουμε και την πρόληψη. Πρέπει και αυτά να χρηματοδοτηθούν. Και το θέμα είναι ποιους μηχανισμούς θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε μερικά βήματα προς τα εμπρός. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν έχει υποβάλει ήδη συγκεκριμένη πρόταση που αφορά το Ταμείο Λιλεγγύης. Θεωρώ ότι το Συμβουλίο και η Κομισιόν έχουν συνταχθεί με την πρόταση της Κομισιόν υπέρ της θέσης δηλαδή που καλεί το Συμβουλίο και τις Προεδρίες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος ο λόγος στην εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα στο τέλος της συζήτησης να σας ε, μιλήσω για τις προθέσεις μου όσον αφορά αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων εσκεμένα δεν θέλησα να επισέλθω σε τεχνικές λεπτομέρειες ή σε συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί αυτό το οποίο θα ήθελα, ήθελα εγώ με αυτή την πρώτη συζήτηση είναι να καταλάβω ποιες είναι οι παράμετροι σύμφωνα με τις οποίες θα προχωρήσουμε στην σύνταξη της γνωμοδότησης. Ήθελα λοιπόν να ε, ακούσω τι απόψει και μέσα από τι παρεμβάσει σα και σα ευχαριστώ για αυτέ, μπόρεσα να καταλάβω σαφώ ποια είναι τα θέματα τα οποία σα απασχολούν περισσότερο. Αυτό το οποίο για μένα ε, είναι ουσιαστική σημασία και ε, έχει να κάνει με αυτά τα δύο επίπεδα προβληματισμού τα οποία ανέπτυξα για προηγουμένω. Πρόληψη και παρέμβαση. Και για άλλη φορά το ξαναλέω. Ο τίτλος μιλά αποκλειστικά για πρόληψη. Ενώ στο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρεται και η παρέμβαση και η διαχείριση. Μπόρεσα λοιπόν με βάση τις παρεμβάσεις να δω ότι υπάρχουν, ότι υπήρξαν συνάδελφοι που αναφέρθηκαν στην πρόληψη, πολύ, ε, στη, στην παρέμβαση. Λίγοι αναφέρθηκαν στην πρόληψη, μόνο, αποκλειστικά δηλαδή μεν ε, για την ε, πρόληψη, η δε για την παρέμβαση, ενώ οι περισσότεροι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν και στα δύο, και στι δύο συνιστώσει. Άρα λοιπόν δεν χωρά αμφιβολία για το ότι οι δύο αυτές συνιστώσει είναι αυτές που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στη γνωμοδότηση. Πρόληψη που σημαίνει ότι βλέπουμε τις αιτίε των φυσικών καταστροφών και των ανθρωπογενών που μπορεί να δράσει ο άνθρωπος και πώς. Γιατί μιλάμε για πρόληψη, ακριβώ αυτό εννοούμε. Πώς μπορούμε να προλάβουμε. Ε, Πρέπει επίση να καταλάβουμε το πώς οι γεωργοί μπορούν να είναι πρωταγωνιστές σε αυτή τη διαδικασία. Πώς με την παρουσία τους, τους αγρούς, στην Ήπεθρο, πώς με τη δραστηριότητά τους μπορούν ε, να προλάβουν τις φυσικές καταστροφές. Και η άλλη συνιστόσα, όταν μιλάμε για ε, παρέμβαση, έχει να κάνει με τις απαραίτητες συνθήκες που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός αυτόματου συστήματος που θα ενεργοποιείται αυτόματα και που θα έχει την απαραίτητη χρηματοδότηση, την επαρκή χρηματοδότηση. Και Βεβαίω όλα αυτά κάτω από την προοπτική της γεωργίας. Παρέμβαση πώς θα είναι αποτελεσματική για να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες των καταστροφών, των φυσικών καταστροφών. Για οι συνέπειες στη γεωργία. Τώρα, ε, όσον αφορά τα φαινόμενα πρέπει να εξετάσουμε. Εγώ ανέφερα πάρα πολλά τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στη γνωμοδότηση. Αλλά βεβαίω είπα ότι θα πρέπει να χαρακτηρίζει η κοινή λογική και θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μα στα φαινόμενα αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερε επιπτώσει στη γεωργία. Πυρκαγιές, ξηρασίες, κυρίω στο νότο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και πλημμύρες στο βορρά. Όσον αφορά κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα, μπόρεσα να δω ότι αναφέρθηκαν τρεις τομείς που φαίνεται ότι έχουν προτεραιότητα. Δασική πολιτική, Βέβαια, εδώ δεν πρέπει να πούμε σε συγκρίσει δάση του νότου, δάση του βορρά. Δεν είναι εκεί το θέμα. Αλλά πρέπει να δούμε και τον χωροταξικό σχεδιασμό, όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν τεράστιε επιπτώσει. Παράδειγμα, πλημμύρε. Όταν υπάρχουν προβλήματα με υπερχείληση των υδάτων, πλημμύρε όπω για παράδειγμα στη Σικελία πριν από ένα μήνα, ε, αυτά έχουν να κάνουν και με τον ε, χωροταξικό σχεδιασμό και με το που βρίσκονται οι οικισμοί των και οι γεωργικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά τα είπα και στην εισαγωγική μου παρατήρηση και, το είπαν και, τα είπαν και οι συνάδελφοι στις, στις ομιλίες τους, στις παρεμβάσεις τους. Αυτά είναι κυκλικά φαινόμενα που εμφανίζονται. Και δεν πρέπει να ε, αποφασίζουμε ε, κάτω από την πίεση των γεγονότων. Πρέπει να αποφασίζουμε νυφάλια και όχι τη στιγμή που ε, προκύπτουν οι φυσικές καταστροφές. Να τα δούμε τα πράγματα με περισσότερη αντικειμενικότητα επίσης, αν δεν βρισκόμαστε κάτω από την πίεση των γεγονότων. με δύο λόγια, νομίζω ότι οι στόχοι που ετέθησαν σε αυτή την ε, πρώτη ε, ανταλλαγή απόψεων επετέφθησαν. Βεβαίω ε, θα σταθώ στα πιο επίγοντα θέματα, στα πιο ευαίσθητα αν θέλετε. Σα ευχαριστώ όλου για τι παρεμβάσει σα και για το γεγονό ότι είπατε ότι είστε έτοιμοι να συνεργαστείτε επικοδομητικά και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. 22-23 Φεβρουαρίου 2010 θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 1η Μαρτίου 2010 και 17 Μαρτίου συνεδρίασή μα θα εγκρίνουμε τη γνωμοδότηση, θα θετήσουμε τη γνωμοδότηση. Ω συνήθω, οι συντονιστέ θα ενημερώσουν ε, την ε, Επιτροπή μας για τα αποτελέσματα τη ε, της του συνεδρίασης. Και βεβαίω είναι η τελευταία μας συνεδρίαση για το 2009. 2006, 2026-27 Ιανουαρίου θα έχουμε την επόμενη συνεδρίαση.